του κυρίου Ντένανο, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την πρόθεση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Έχετε τον λόγο. Αλλά, πρώτα απ' όλα, ε, να σας πω ότι έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή που φοβόμαστε για μια κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ε, με σοβαρές ε, επιπτώσεις προς το γεωργικό τομέα, θα σας παρουσιάσω ένα κλάδο που είναι σημαντικό διακύβευμα για την ε, μελλοντική μας επιστημιστική ασφάλεια. Ε, είτε καταναλώνουμε άμεσα μπιζέλια ή προϊόντα με βάση τη είτε τα χρησιμοποιούμε για τις ζωοτροφές, τα, οι πρωτενούχες καριέργειες βρίσκονται στο κέντρο της ε, ε, διατροφής μας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τα συστήματα υφόρου παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αξιοποιήσουμε τις καλλιέργειε αυτές και να θαρρύνουμε τους ε, γεωργούς να ασχοληθούν με αυτή την καλλιέργεια για να ενισχύσουμε επίση την ανταγωνιστικότητά του. θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι είδου γεωργία θέλουμε για το μέλλον και τι είδου πρότυπου διατροφή σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό, η υπογραφή των συμφωνιών GATT και Blair House ε, και η σταδιακή, το σταδιακό άνοιγμα των αγορών σφράγγισε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσμα σήμερα εισάγουμε το 75% των φυτικών πρωτεϊνών από την Αργεντινή, τη ΣΥΠΑ και τη Βραζιλία με όλο και μεγαλύτερη αύξηση του ελλείμματό μας. Και μάλιστα ενώ η Κίνα έχει εφαρμόσει στρατηγική εφαρμογή ε, ε, ανεφοδιασμού με συμβάσεις παραγωγή αδιαφανής, ε, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, εμείς ε, αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση και πρόβλημα λόγω της σταθερότητας των αγορών. Και φυσικά να μην ξεχνούμε και την αποψήλωση και το τεράστιο αποτύπωμα του άνθρακα των εισαγωγών μας σε φυτικές πρωτεΐνες. Μάλιστα έχουμε και τις απαιτήσει των Ευρωπαίων πολιτών που θέλουν όλο και λιγότερα προϊόντα με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα προϊόντα σόγιας είναι γενετικώς τροποποιημένα. Ε, επίσης, ε, ε, έχουμε μεγάλες απαιτήσεις. Μήπως όμως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον, στην κτηνοτροφία μας που χαρακτηρίζεται από ποιότητα και χνηλασιμότητα και θα απειληθεί λόγω αυτής της εξάρτησης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οι γεωργοί, οι οργανώσεις, η παραγωγή τροφίμων, οι ερευνητές, οι διοικήσει και οι βουλευτές να συνεργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική κάτι πολύ αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εφοδιαστούμε με ένα ουσιαστικό σχέδιο στρατηγικού ενεφοδιασμού ε, με έμφαση στην έρευνα και στην, ε, στο εμπόριο με βραχία λυσίδα ενεφοδιασμού. Θα πρέπει επίσης να μειώσουμε την πίεση εδάφη και τα δάση της ε, Λατινικής Αμερικής και αυτός ο αγώνας κατά της αποψήλωσης των δασών βρίσκεται στην καρδιά και του των συμφωνιών του Παρισιού για το κλίμα. Αλλά δεν θα έχουμε αύξηση της παραγωγής αν δεν βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα αυτών των καλλιεργιών. Σήμερα η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών είναι πολύ λιγότερο αποδοτική από τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Ε, δεν θα πρέπει να μπορούμε που μόνο 3% των αρρώσιμων καλλιεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορούν πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Βέβαια, τα ψυχανθή έχουν τεράστια αποτελέσματα πλεονεκτήματα. Ε, δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και περιορίζουν τη χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων. Επίσης, ε, συμβάλλουν στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντάσσονται στην κυκλική οικονομία. Ε, τα γεωπονικά πλεονεκτήματα των αζωτοδεσμευτικών φυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ΚΑΠ μαζί με την σπορά, τη συγκαλλιέργεια και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στις πρωτεϊνόχες καλλιέργειες, αλλά και στα, κτηνιατρικά, στα κτηνοτροφικά συγγνώμη, φυτά και τη χορτονομή που είναι η σημαντικότερη πάροχη πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Επίση, μια καλύτερη εδαφική διάρθρωση του κλάδου διεκδικούμε. Θα ήθελα να έχουμε και συνδεδεμένε ενισχύσει, ώστε να μπορέσει ε, η γεωργία μα να στραφεί στην καλλιέργεια ψυχανθών. Ε, επιστηστική ασφάλεια, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, κύκλος του αζότου, όλα και η παραγωγή των πρωτεϊνών είναι σημαντικά διακυβεύματα της μελλοντικής μας γεωρικής πολιτικής. Γι' αυτό και θα πρέπει η μελλοντική ΚΑΠΑ να αναδείξει την αξία των πρωτεϊνικών καλλιεργειών. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές και όλους τους συνεργάτες μου που μου επέτρεψαν να εκπονήσω την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στην διαδικασία και έτσι αλλά σήμερα πρέπει να ολοκληρώσουμε ακριβώς στις 11 η ώρα. Τρεις ε, συναδελφοί από το ΕΛΚ. Ακούσατε τα ονόματα. Ο κύριος ε, Φάντα Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αυτοί οι συνάδελφοι, η στρατηγική για τις πρωτεΐνες έχει μεγάλη σημασία. Και στην ε, Ευρώπη τη δεκαετία του 90 απαγορεύσαμε τις ε, ζωικές πρωτεΐνες στις ε, ζωοτροφές ε, και δικαίως. Αυτό σημαίνει ότι εισάγουμε μαζικά σόγια από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Πρέπει να περιοριστεί αυτή η εξάρτηση και να προωθήσουμε άλλες ε, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Αλλά πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και άλλες πηγές πρωτεϊνών. Από φύκια παραδείγματος χάρη από έντομα. αυτά έντομα όμως απαγορεύονται από την δεκαετία του 1990 και αυτό ζητάω από την Κομισιόν να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την δυναμική των εντόμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντζιου για ένα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω να συγχαρώ και να ποτίσω φόρο τιμής ε, στο συνάδελφο Ζαν Πολ για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ψέματα ε, στους εαυτούς μας. η παραγωγή ψυχανθών και προϊόντων σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική ε, και κυρίως ε, σε μεγάλο βαθμό έρχεται από το εξωτερικό, ιδίως για τη σόγια και μάλιστα η σόγια είναι γενετικώς τροποποιημένη. Έτσι είναι η πραγματικότητα και κανένας δεν το λέει, παρά το γεγονός ότι οι γενετικώς τροποποιημένες ε, καλλιέργειες απαγορεύονται στην Ευρώπη. Πρέπει να ε, υπάρχει ένα σχέδιο πρωτεουνούχων ε, καλλιεργειών στην Ευρώπη και να έχουμε πλήσιε πρωτενε χωρί γενετικώ τροποποιημένε οργανισμού, κυρίω στη σόγια, και να ε, μην χρειάζεται να ε, ε, έρχονται από το εξωτερικό. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να εντοχθεί αυτό το σχέδιο για τις πρωτεΐνες στην ΚΑΠ μετά το 2020 και να βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου Ντενανό θίγει πραγματικά το σοβαρό ζήτημα της επισητιστικής ασφάλειας διότι έχει αποδειχθεί ότι οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και οι καλλιέργειες ψυχαρθών φυτών δεν έχουν αναπτυχθεί όσο έπρεπε στην ευρωπαϊκή ένωση. το 35% από όλα αυτά τα φυτά και τις αντίστοιχες ουσίες εισάγονται στην ευρωπαϊκή ένωση και σίγουρα η σόγια που εισάγεται από τις ηνωμένες η οποία είναι γενετικώς τροποποιημένη και γι' αυτό το λόγο ορθώς υπάρχει μια τεράστια αντίδραση και από το ευρωκοινοβούλιο αλλά φυσικά και από τους ίδιους τους καταναλωτές η κίνα ταυτόχρονα χρησιμοποιεί μια διαφορετική στρατηγική έχει συνάψει μια αποκλειστική ουσιαστικά αδιαφανή συμφωνία με τη βραζιλία έχει επενδύσει σε υποδομές παραγωγής σε λιμενικές μεταφορές και με αυτόν τον τρόπο ανταγωνίζεται θα έλεγα και σε μεγάλο βαθμό αθέμητα την ευρωπαϊκή ένωση. πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτάσεις της έκθεσης του συναδέλφου denanot. ευχαριστώ. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τον συνάδελφο τον Ανώ, τον οποίο συγχαίρω για το έργο του, είχα την αίσθηση ότι γυρίσαμε πίσω στο χρόνο, πριν από μία ευθετία, όταν συζητούσαμε την έκθεση Χόισλινγκ. Οι ίδιοι λόγοι, οι ίδιοι όροι, η ίδια ίδια διατύπωση, ίδιες ελπίδες, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει. Ε, έχουμε τεράστια εξάρτηση στην εισαγωγή πρωτεϊνών και 20, έλλειμμα 20 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφών. Και στην ΚΑΠ έχουμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, αλλά χρειάζεται πρώτα απ' όλα κάποια συνοχή, κάποια συνέπεια. Και οι προτάσεις του 2017 για τις περιοχές οικολογικής εστίασης έχουν μια μικρή επιρροή στις καλλιέργειες ψυχανθών. Επίσης, ε, λαμβάνονται υπόψη και τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας, γιατί οι πλακούντες σόγιας και άλλων κτηνοτροφικών φυτών χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές, ε, αλλά επειδή πολλές πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα δεν έχουμε τόση σημαντική αξιοποίησή τους για τις ζωοτροφές. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς αν θέλουμε πραγματικά να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Ο κύριος Μπούντα. Μια μεγάλη πρόκληση για την γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφαλής παροχή πρωτεϊνών και βεβαίως και για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος και για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα πρωτεϊνούχα φυτά είναι πολύ σημαντικός πόρος και για το περιβάλλον. Γιατί δεσμεύουν και το άζωτο βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους και δημιουργούν καλές συνθήκες για την βιολογική καλλιέργεια. Γι' αυτό ακριβώς ε, το εθελοντικό πρασίνισμα του δεύτερου πυλώνα πρέπει να λάβει υπόψη την ε, ευελιξία και την στήριξη για τις ε, πρωτεϊνούχες ε, τροφές και να υπάρχει οικονομική στήριξη και μετά το 2020 χρειάζεται μια δική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Να σας πω όμως πόσο σημαντικό είναι να έχουμε νέα μέσα στήριξης για τα πρωτεϊνούχα που μπορούν να αφαιρεθούν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως επίσης και το κόκκινο τριφύλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Πόλτσακ είναι ο τελευταίος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατά την απόψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να πω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει εξαρτημένη από τις διάφορες εισαγωγές. Ε, ιδιαίτερος όταν ε, στην συγκεκριμένη περιοχή έχει πλέον η Κίνα το πάνω χέρι. Πρέπει να είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα φυτά ή να έχουμε αξιόπιστες χώρες από τις οποίες να μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Ε, προσωπικά εγώ στηρίζω την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές της Αϊφόρου ή μια συμφωνία με την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οι τρεις βουλευτές που ήθελαν να μιλήσουν θα λάβουν τον λόγο, αλλά Δεν θα να τον λόγο στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, κύριε Πετήρη, έχει τον λόγο τώρα. Ε, κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της ανεπάρκειας φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ε, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση πρωτεϊνικών καλλιεργειών, γιατί δυστυχώς σήμερα εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι οι περισσότερες τροπολογίες οι δικέ μου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο έγιναν δεκτέ από τον εισηγητή. Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών στις γεωργικέ εκτάσεις είναι σημαντικό μήνυμα και γι' αυτό θα πρέπει και στις αεροτρές καλλιέργειες αλλά και στα κτηνοτροφικά φυτά να προωθούμε τις ε, πρωτεϊνικές καλλιέργειες ε, όπως τις όγιας, κουκιών, μπιζελιών καθώς και τριφυλιού και πολλών ψυχανθών. Είναι σημαντικό κάτι τέτοιο. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις, περιφερειακούς, τις περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής τις, ε, για, την, και, για την παραγωγή και επεξεργασία των πρωτεϊνών και την οργάνωση των γεωργών καθώς και τη συνεργασία γεωργών και κτηνοτρόφων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να προωθήσουμε ε, τι ε, τις ενισχύσεις της ΚΑΠΑ για την προώθηση των, ψηφι, Χαιρετίζω τον ενδιαφέρον των, ε, των, καταναλωτών για προϊόντα χωρίς γενετικώς τροπημένες οργανισμούς και τις πρωτοβουλίες αντισόγια δούναβη που εξασφαλίζουν ποιοτικά πρωτεϊνούχα προϊόντα. Ο Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ζητήσω το λόγο στο επόμενο ΚΑΤΣΤΙΑΗ σε καμία συζήτηση από εδώ και πέρα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο κύριος Ντενανό, οι μας, έκανε μια εξαιρετική παρέμβαση. Ε, μίλησε για την κατάσταση στην Ευρώπη, την οποία ανεχτήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και από ε, τη μια προσπαθούμε να είμαστε πολύ ιδεολόγοι και από την άλλη προκαλούμε περισσότερη ζημιά. Ε, είπαμε για εισαγωγές, εμείς δεν θέλουμε γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και τελικά είναι γενετικώς τροποποιημένα αυτά που εισάγονται. Επίσης, το αποτύπωμα του άνθρακα πρέπει να ε, είναι πολύ πιο λογικό να παράγουμε εδώ στην Ευρώπη και να έχουμε και ωφέλη για τους ε, γεωργούς μας. Και επίσης όπως ε, τονίστηκαν υπάρχουν και πρόσθετα ωφέλη. Για παράδειγμα, μείωση του αζότου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ ήμουν εισηγήτης για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπήρχε μια πρόταση να σταματήσει να χρησιμοποιείται αυτή η εισαγωγή. Ευτυχώς το Κοινοβούλιο ε, ε, προτείνει να προωθήσουμε τις καλλιέργειες εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέντα. Έχετε το λόγο. Α, δεν θέλετε το λόγο. Εντάξει, το διαγράφουμε το όνομα από τον κατάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο λοιπόν έχει τώρα για λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον κύριο Ντενανό, για την προετοιμασία αυτή τη έκθεση ίδια πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση των Πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Οι προκλήσεις και ευκαιρίε ε, που αντιμετωπίζει ο πρωτεϊνικός ε, τομέας των καλλιεργιών και το ενδιαφέρον ε, των ενδιαφερομένων αναφέρονται σαφέστατα σε αυτή την έκθεση. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι πρωτεϊνικές καλλιέργειες είναι σημαντικές ε, για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία ως αναπόσπαστο τμήμα των ζωοτροφών και πηγή αμινοξέων για, τις, για, τα, για τα ζώα και γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς ε, στην ε, ε, κατανάλωση των ανθρώπων. Και η πρωτεϊνική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα βοηθήσει και τους γεωργούς και τους ε, παραγωγούς ζωοτροφών και θα παρέχει τρόφιμα και για τους καταναλωτές, αλλά θα συμβάλλει και σε έναν μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών και κλιματικών ωφέλων. Για παράδειγμα, η δυνατότητα να ε, μειώσουμε την περιεκτικότητα ζώτου στην ατμόσφαιρα. Υπό αυτή την έννοια, η έκθεση ίδια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτη και συμβάλλει πολύ στην προετοιμασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σχέδιο για τι πρωτενε, το οποίο προγραμματίζεται για δημοσίευση μέχρι το τέλο του έτου. Αυτή η δημοσίευση θα ε, συνοδεύεται και από μία ε, ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τις ε, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες το Νοέμβριο στη Βιέννη, στη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου και θα ήθελα να τονίσω και το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η μελλοντική Αυστριακή Προεδρία σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Η ε, πρωτεϊνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχο έχει να παρέχει βιώσιμη παροχή πρωτεϊνών, λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτάρκης μόνο κατά 38% για την ε, βασική πηγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών και ε, μόνο 45% επάρκεια για τους ε, φλακούντες σόγιας που είναι και βασική και πολύ σημαντική πηγή πρωτεϊνών. Γι' αυτό εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή σόγιας που έχει και σημαντικές ε, παγκόσμιες συνέπειες. Μία μελέτη που έγινε το 2013 ε, διαπίστωσε ότι η επέκταση της σόγιας είναι υπεύθυνη για το 19% ε, της παγκόσμιας αποψήλωσης μεταξύ του 1990 και του 2008 κυρίως στη Λατινική Αμερική. Επίσης υπάρχουν και διάφοροι πρακτικοί λόγοι που εξηγούν γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα και δεν αντιμετωπίζεται τόσο εύκολα. Αυτό περιλαμβάνει τις αγρονομικές συνθήκες στην Ευρώπη, την οικονομική ε, δυνατότητα που προσφέρουν αυτές οι καλλιέργειες ε, και το, ε, τις επιδοτήσεις σε σχέση με τις εισαγωγές και διεθνείς δεσμεύσει στον ΠΟΕ που μειώνουν το ε, επίπεδο στήριξης για ε, παραγωγή ελαιούχων σπόρων. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μια λύση πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το πεδίο εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τις Πρωτεΐνες λοιπόν θα είναι ευρύτατο, θα παρέχει όλες τις ε, χώριες πηγές ε, για παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών, καθώς επίσης και τη ζήτηση που υπάρχει. Ε, σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το ευρωπαϊκό σχέδιο λοιπόν θα επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς ε, που τονίζονται και αυτοί στην έκθεση του κύριου Ντενανό. Έρευνα και καινοτομία για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όσον αφορά τη βελτίωση των ειδών και καλύτερη προσαρμογή σε κλιματικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγρονομικά ωφέλη των πρωτεϊνικών καλλιεργιών, καθώς επίσης ε, διαφορές πηγές προμήθειας και αλυσίδα αξιών, καθώς επίσης και δυνατότητες στην αγορά για, τα, ε, για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες σε διάφορες τομείς αγοράς. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται και στην σημασία της στήριξης μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής για την παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών. Πράγματι, η κοινή γεωργική πολιτική παρέχει μια σειρά από μέτρα τα οποία είτε έμεσα ούτε άμεσα ε, ενθαρρύνουν την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Οι συζητήσει εν εξελίξη για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα ε, δώσουν και τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε περαιτέρω τη στήριξη μέσω πολιτικής για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Η έκθεση του Κοινοβουλίου τονίζει επίσης και τη σημασία του ερευνητικού έργου, το οποίο ε, θα βρίσκεται μεταξύ των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρώτη γραμμή. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη αυτού του σχεδίου για τις πρωτεΐνες, το οποίο θα είναι προ όφελο όλων εν τέλει, διότι η Ευρώπη θα είναι περισσότερο αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή των ουσιαστικών πρωτεϊνών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε.